Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε αυτή την συνεδρίαση για το πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων. Έγκριση της ημερήσια διάταξης, εγκρίνεται. Δεν έχουμε ανακοινώσει στο σημείο 2. Και έτσι λοιπόν περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης για την ε, για την δημιουργία του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Θα, θα πρέπει να το δώσουμε πραγματικά στις 16 και 45 να σας ενημερώσω και πραγματικά θα πρέπει να σεβαστούμε τα χρονικά όρια. Χρόνος αγόρευσης λοιπόν και ξέρετε ότι θα είμαι αυστηρός με το χρόνο ομιλία σας, αν δεν το πράξετε εσείς δηλαδή. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους δύο συνεισηγητές για τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά εκαστός από την Επιτροπή Προεπιλογισμών Κταρχάς, Σοσιαλδημοκράτες, Γκάρδια Ζαβάλ Ρουμπιάλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό των τεσσάρων λεπτών. Επιτέλους, έχουμε την πρόταση σχεδίου του προεπολογισμού, αλλά ε, όχι όπως την τελευταία φορά που δεν την είχαμε, δεν βρεθήκαμε, συζητήσαμε πάρα πολύ, συνεισηγήτρια και εγώ και τελικά καταφέρουμε να καταλήξουμε μια συμφωνία και ε, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία θα τα μεταθέσουμε για την επόμενη φάση, τη φάση των τροπολογιών πάντως. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμφωνίες και τελικά έχουμε 51 τροπολογίες επί της πρότασης της Επιτροπής. Έπρεπε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για τους στόχους του προγράμματος. Και επίσης θα πρέπει να γίνει και ευθυγράμμιση για όσο αποφασίσαμε και ψηφίσαμε για το ΠΔΠ, όσα είπαμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπότε και συνδέθηκε στο θέμα με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους στόχους, τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού και είπαμε ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν και οι χώρες εκτός ευρώ για την απάτη, προβλέπονται δράσεις, την δίκαιη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και αυτό άλλες τροπολογίες, δέσμη τροπολογιών είναι αυτά που αφορούν την μεταρρύθμιση των κρατών μελών. Και εδώ είπαμε ότι έχουμε μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προτείνουν αντισταθμιστικά μέτρα για τις τυχόν αρνητικές συνέπειες της μεταρρύθμισης. Οι δε αεφορολογικές αρχές θα πρέπει να ασχοληθούν με τα δημοσιονομική πλευρά αυτών των μεταρρυθμίσεων. Πιστεύω ότι θα τελειώσουμε στο χρονοδιάγραμμα, αποκλείσαμε την πιθανότητα του να μεταφέρουν εδώ πόρους ε, οι δημοσιομικές αρχές από άλλα προγράμματα προς αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Τίποτα άλλο και θα συστήσουν ξανά αυτά που βρίσκονται επί της τραπέζης. Ο Πρόεδρος. Έντερ, ευχαριστούμε. Η κυρία Νάκτικαλ που είναι η Καρολίνη, η συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ. Υποστηρίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα υποστηρίξης των μεταρρυθμίσεων για την ε, ενίσχυση της ανάπτυξης και της οικονομικής ανθεκτικότητας της Ένωσης. Αυτό θα κάνει την Ένωση πιο ισχυρή, θεωρώ, και θα απαλύνει και τις αρνητικές επιπτώσεις των μελλοντικών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ολοκληρώσαμε το σχέδιο έκθεσης η συνεργασία μας πάει πάρα πολύ καλά, είναι με καλό πνεύμα, αλλά φαντάζομαι ότι σε τελική ανάλυση θα υπάρχουν ιδεολογικά κενά τα οποία θα πρέπει να γεφυρώσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν συμπερέσνουμε, μάλλον συνάψαμε ένα σχέδιο συμβιβασμού σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή των θεσμικών οργάνων της Ευρωζώνης και διάφορες προτάσεις σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Ένας από τους στόχους μου λοιπόν ήταν να να ενισχυθούν οι ισολογισμοί και σε ό,τι αφορά το είδος των μεταρρυθμίσεων που θα πρέπει να δικαιούνται ε, η οικονομική ενίσχυση και φυσικά η ευθύνη είναι στα χέρια της Επιτροπής σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τις συστάσεις αναχώρα, αξιολόγηση της πρότασης και τελικά εκτίμηση για το αν θα πρέπει να καταβληθεί η πληρωμή. Η διαδικασία λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει, να έχει πιο, πολύ, πιο πολλές δικλείδες ασφαλείας και χαίρομαι που καταφέραμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Επίσης προτείνεται τα ανεξάρτητα όργανα εποπτείας που έχουν συσταθεί στα κράτη-μέλη να μπορούν και αυτά να προτείνουν προτάσεις για τις δεσμεύσεις. Ένα Μία αξιολόγηση από ανεξάρτητο σώμα θεωρώ ότι θα βοηθήσει και τα κρατημέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δεύτερη, το δεύτερο επίταγμα είναι ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε για το παιδί εφαρμογή για την υπηρεσία αυτή. Μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις για να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στι συνθήκε. και θα πρέπει να τηρούνται και οι σχετικέ νομοθεσίε στην Ευρωζώνη. Τρίτον, συμφωνήσαμε για τη βελτίωση τη πρόταση σε ό,τι αφορά τι δεσμεύσει ε, μεταρρυθμίσεων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξηγήσουν λοιπόν ποιε μεταρρυθμίσει έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τι προτινόμενε μεταρρυθμίσει. Οι διατάξει αυτέ θα βελτιώσουν ε, τη βάση της απόφασης ε, που έχει ληφθεί από την Επιτροπή κάποια από τα πράγματα για τα οποία δεν συμφωνήσαμε τώρα και γι' αυτό και το τμήμα αυτό έμεινε εκτό του σχεδίου έκθεση. Καταρχά, τη φορά το πεδίο εφαρμογή του προγράμματο. Για μένα είναι κρίσιμο η οικονομική ενίσχυση να δίδεται σε αντιρφωτικέ μεταλλεκμήσει που θα συμβάλλουν στην οικονομική άντοχη των κρατών μελών και τη Ένωση. Και γι' αυτό η σαφή ε, σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τι συστάσεις αναχώρα θα πρέπει να ιδρυθεί όπω προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην σα πω και να ενισχυθεί. Η διάβρυνση του πεδίου εφαρμογή θα συνεπάγεται ηθικό κίνδυνο. Αυτό είναι μεγάλο κίνδυνο. Χρειάζονται λοιπόν αυστηρά κριτηρία για την επίτευξη των στόχων. Δεύτερον, δεν συμπεριλαμβάναμε αναφορά στο κράτο δικαίου στο σχέδιο έκθεση μια και Όλοι θέλουμε σαφή αιρεσιμότητα στι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίσαμε να καταθέσουμε χωριστά λοιπόν τι τρολογίε αυτέ. Και είναι σαφέ για μένα ότι κανένα κράτο μέλο δεν θα είναι επιλέξιμο αν δεν εφαρμόζει τι κοινέ μα αξίε. Τελευταίο σημείο, ο συντελεστή για την κατανομή των κονδυλίων. Ευαίσθητο σημείο Μια και θα σημαίνει αυτό κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, δίδοντα όμω και μεγάλα κίνητρα για τα μεγάλα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι το σχέδιο έκθεση αποτελεί μια καλή βάση για τι μελλοντικέ μα συζητήσει. Προσβλέπω στις τροπολογίε καθώ και στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Ναχτχαλέη, ο πρόεδρο, και στη συνέχεια να ακούσουμε από δύο λεπτά του σκιώδει. Ο κ. Λαμάσορ από το ΕΛΚ, από την Επιτροπή Προπολογισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, εν ονόματι του ΕΛΚ για την Επιτροπή Προπολογισμών. Συγχαρητήρια στην κυρία Κατήσια Μπάλ για την έκθεσή τη. Κάποια σχόλια ή ερωτήσει. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση. Είναι ο μηχανισμός στήριξης της σύγκλησης. Εγώ ε, θα ήθελα να αυξήσουμε το μερτικό που πάει σε αυτό το μηχανισμό. Ούτω ώστε οι χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη να κάνουν τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει για να μπουν στην Ευρωζώνη. 20% των συνολικών πιστώσεων προτείνω να μπουν σε αυτή τη δράση. Για το υπολογισμό τη οικονομική τη μέγιστη συνεισφορά, ένα μόνο κριτήριο είναι ο αριθμό των κατοίκων και είναι κάπω παράδοξο στοιχείο και προτείνω να συνδυαστεί το κριτήριο του πληθυσμού με αυτό του εισοδήματος, κατά κεφαλή. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων, πολύ ευαίσθητο θέμα πολιτικά, πρέπει να αποφευχθεί. Οι μεταρρυθμίσεις θα διαρκήσουν πολλά χρόνια. Αλλαγέ πλειοψηφιών ε, και κυβερνήσεων γίνεται μετά από τις δημοκρατικές εκλογές και οι δημοκρατικές χώρες που είναι δικαιούχοι αυτών των ε, μέτρων αλλάζουν τις μεταρρυθμίσεις. Αντί να αλλάξει η προθεσμία, η περίοδος η πενταετής, προτείνω μια, να υποβάλλεται σε πολιτικό έλεγχο ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων. Και ο έλεγχος ξεπερνά τα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να προσφύγουμε σε ένα σύστημα αντίστροφης πλειοψηφίας στο Συμβούλιο συγκρίσιμο με αυτό που ισχύει στο six pack και στο two pack. Όσον αφορά την αρεσιμότητα στην εκλογική σκέψη 46, η καλύτερη λύση θα ήταν μια οριζόντια ρήτρα για όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Επιτροπή Προπολογισμών προς αυτή την κατεύθυνση κατευθύνεται. Και τέλος, διερωτώ με, η δημιουργία of Independent Fiscal Institution, τι νόημα έχει. Έχουμε ήδη τέτοιους φορείς σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμασούρ. Η κυρία Μάλετιτς ε, για το ΕΛΚ, για την ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Η κατανομή δεν μπορεί να βασίζεται στον αριθμό των πολιτών και θα πρέπει να δούμε πώς η διαδικασία θα είναι και απλή, λαμβάνοντας όμως υπόψη τον περίπλοκο χαρακτήρα των προσεφαρμογή μεταρρυθμίσεων, βάσει των αναχώρα συστάσεων και διάφορες μακροοικονομικές ανισορροπίες να ληφθούν υπόψη. Και όπως συνάδελφος Λαμασούρ είπε, και το επίπεδο ανάπτυξης να λαμβάνεται υπόψη. ΑΕΠ σαν ποσοστό του μέσου όρου του ΑΕΠ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Δεν μπορούμε να διαθέσουμε ε, το μισό ποσό στην ανταγωνιστικότητα. Χρειαζόμαστε λίγα περισσότερα για αυτή την πρώτη φάση και πρέπει να ισχύει για το, το πρώτο εικοσάμινο των δαπανών. Για τον εξάρτητο ε, δημοσιονομικό φορέα δεν είμαι αρνητική, αλλά δεν μπορεί να σχετιστεί με τον κανονισμό. 473-2013 διότι αυτό αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μόνο και πρέπει να ακολουθήσουμε πιο ευρεία προσέγγιση όσον αφορά την έννοια. Να διαγράψουμε τα τμήματα που αφορούν τις μεταφορές ε, που είναι υπό κοινή διαχείριση, οι πόροι αυτοί, να πάνε στο κοινό πρόγραμμα και θα πρέπει όμως να υπάρχει συντονισμός των επενδύσεων από την πολιτική συνοχής που σχετίζεται με τις εκθέσεις αναχώρα και μακροοικονομικές ρεσιμότητες και δράσεις που περιλαμβάνονται στις υποχρώσεις προς μεταρρύθμιση που έχουν υποβάλει από τα κράτη-μέλη για να τύχουν υποστήριξη στα πλαίσια του εργαλείου της μεταρρυθμίσης και στους γενικούς και ειδικού στόχους να βάλουμε να ε, υπάρξει μια αλλαγή στον τομέα το δικαστικό και στα συνταξιδοτικά. Ευχαριστώ για το δίλεπτο που τηρήσατε. Σοσιαλιστές ο κ. Μαυρίδης δεν είναι εδώ, εκ μέρους Πάμε στο ECR. Θα πάρετε το λόγο εσείς. Ορίστε. Ευχαριστώ. Εν ονόματι του συναδέλφου του Κώστα Μαυρίδης που ζητά συγγνώμη που απουσιάζει να αναφέρω πέντε σημεία θέλω που ήθελα να αναφέρει εκείνο. Δέχεται ευνοϊκά την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής που εδράζεται επί προγράμματος υφισταμένου. Επιμένει όμως επί κάποιων μαθημάτων πρέπει να αντλήσουμε επί των όρων εφαρμογής και υλοποίησης των προγραμμάτων. Το πρώτο, μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2008, καθένας λαμβάνει υπόψη τη σημασία που έχει η σύγκληση οικονομική και κοινωνική και ανάγκη που υπάρχει να διορθωθούν τα δύο αυτά στοιχεία διορθώνοντας τις αρνητικές πτυχές των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που είναι υπερβολικά εκτεταμένες και να μπορέσουν οι πολίτες να βελτιώσουν το, τη διαβίωσή τους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη δηλαδή ταυτόχρονα τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και να υπάρχει και ευθυγράμμιση με τους αναπτυξιακούς στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη που συμβαίνεται σε τέτοια μεταρρύθμιση. Δεύτερον, ανησυχεί για το πώς τέτοιες μεταρρυθμίσεις θεωρούνται από πλευράς πρικοδότησης από τα κράτη-μέλη, διότι το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν φαίνεται να είναι το μόνο σχετικό πλαίσιο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να κάνουν μεταρρυθμίσεις εκτός του εν λόγω πλαίσιου. Τρίτη παρατήρηση θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσει θα πρέπει να είναι τέτοιε ώστε να αυξήσουν την ποιότητα απασχόλησης, των θέσεων απασχόληση, να αυξηθούν σε απασχόληση, η εθική συνοχή, καταπολεμηθεί η φτώχεια, να υπάρχει σωστός και δίκαιος ανταγωνισμός. Γι' αυτό η σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν είναι κάτι επαρκές και θα πρέπει κάθε μεταρρύθμιση να συνοδεύεται από την εφαρμογή του άρθρου 9 των συνθήκων, το οποίο απαιτεί ανάλυση κοινωνικών επιπτώσεων πριν την πραγματοποίηση κάποιας μεταρρύθμισης. Τέταρτο σημείο, ανησυχεί μήπως ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να μειώσει ε, την πολιτική συνοχή, την πρικοδότηση πολιτική συνοχή να οδηγήσει σε μια ρησιμότητα μακροοικονομική, κάτι που θα έχει αρνητικέ συνέπειε και για τι χώρε που ακόμα έχουν να υποστούν τις συνέπειες των δημοσιονομικών πολιτικών, των σκληρών. Θα πρέπει ο καθένας να πλησιάσει το θέμα με υπευθυνότητα και επικοδομητικά και αυτό θα κάνει από την πλευρά του. Ευχαριστώ πολύ. το SR. Ο κ. Γκέλμερ έχει το λόγο. Για δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αυτό το κοινοβούλιο συμφωνεί επί τη αρχή όταν μιλάμε για θέματα προπολογισμού ότι χρειαζόμαστε πιο πολλή διαφάνεια, πιο πολλή σαφήνεια και πιο πολύ καταμέτρηση τη αποτελεσματικότητα. Άρα δεν καταλαβαίνω από τελευταία... τον τελευταίο καιρό μιλάμε για νέα προγράμματα τα οποία θέλουμε να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι αντίθετα από την διαφάνεια, αδιαφάνεια. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί πέρα από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η πολιτική συνοχή σε εδώ και καιρό, θέλουμε να δημιουργήσουμε μόνιμα προγράμματα. Αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, η πολιτική συνοχή είναι το καταξοχήν εργαλείο αλλά στην πολιτική συνοχή θα πρέπει να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Να καταμετρήσουμε λοιπόν την ε, αποτελεσματικότητα. Δεν μπορούμε απλά να δίνουμε πόρους και κονδύλια και να λέμε εντάξει κάποιο τόπο θα πιάσουν. Δεν είναι λοιπόν να τα συμφωνήσουμε όλα αυτά. Ένα άλλο στοιχείο που καλύπτεται στην έκθεση αυτή γιατί συνέχεια γίνεται μία σύνδεση και αναφορά στην Ευρωζώνη. Όταν λοιπόν έχω ένα πρόγραμμα για την Ευρωζώνη, δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί μιλάμε για υψηλά ποσά εδώ, αλλά δεν μιλάμε για ποσά τα οποία θα χρειάζονταν για να καταστήσουν βιώσιμη την Ευρωζώνη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και να παραδεχτούμε με αφήνει ότι το ευρώ έχει καταρρεύσει, έχει αποτύχει και λοιπόν πρέπει να καταρχίσουμε την Ευρωζώνη γιατί δεν πρόκειται να ανακλητώσουμε τέτοια ποσά. Ευχαριστώ πολύ. Και για να πετύχουμε πραγματικά στερεοφωνική εμπειρία θα δώσω το λόγο και από την στο στην Ευχαριστώ πολύ και να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, οι οποίοι θεωρώ ότι κατέβαλαν πάρα πολλές προσπάθειες για να καλύψουν τα κενά που τους καλύπτουν και τις διαφορές που έχουν στην έκθεση αυτή. Έχουμε και βατικά και αρνητικά να σημειώσουμε. Καταρχάς, στα αρνητικά. Πιστεύω ότι θεωρώ ότι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά το θέμα του ηθικού κινδύνου και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου κράτη τα οποία δεν έκαναν εγκαίρως τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που τους αναλογούσαν, τώρα ε, θα μπορούσαν να έχουν ε, σημαντικές ε, οικονομικές επιδοτήσεις. Αυτό προφανώς δημιουργεί κίνητρο, λάθος κίνητρο. Ή θα μπορούσε, εν περιπτώσει, να δώσει λάθος κίνητρα, να μην κάνουμε λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις και βλέπουμε μήπως μας δώσουν και χρήματα για τις καθυστερισμένες αυτές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να το επιτρέψουμε αυτό. Χρειάζονται μηχανισμοί ασφάλειας για να το αποτρέψουν αυτό, για να μην υπάρξει εσφαλμένη τέτοιο κίνητρο. Και δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά δυστυχώ τέτοιο μηχανισμό ασφάλεια. Και επίση και το front loading αποτελεί πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν αυτές οι επιδοτήσεις, κατά πόσον μπορούμε να δώσουμε επιδοτήσεις για μεταρρυθμίσεις που δεν χρειάζονται οποιαδήποτε επένδυση. Σταθετικά τώρα. Να σημειώσουμε τον ανεξάρτητο οργανισμό που δημιουργείται. Σωστό βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αν και δεν επαρκεί για την καλή μεταρρύθμιση και εφαρμογή του προγράμματος. Και τέλος, μια παρατηρήση για την πολιτική συνοχής και αυτό που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, η νομική βάση είναι η πολιτική συνοχή και να σας επιθυμίσουμε ότι η πολιτική συνοχή ε, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. άρθρα 174 της Συνθήκης. Εδώ όμως μπαίνει στο επίκεντρο η Ευρωζώνη. Και υπάρχουν και δύο μέλη τα οποία δεν θα είναι στην Ευρωζώνη και άρα δεν μπορούμε να αναφέρουμε εδώ την Ευρωζώνη και ενδεχομένως λοιπόν να μην έχουμε καν νομική βάση στην παρούσα φάση. Although we don't seem to have anyone from the budgets committee. So, um, from um, the Greens, Mr. Από τους πράσινους ο κ. Γκίγκολ δεν είναι εδώ. Ο κ. Λάμπερτς, μήπως θέλει να πει τίποτα. Είμαι ο μόνος πράσινος. Έχω τα τέσσερα λεπτά όλων των πρασίνων. Τρία λεπτά. Πώς σας φαίνονται τρία λεπτά. Είμαι, δεν είμαι σκιώδης. Για κανέναν από τους συνεισηγητές, αλλά μου ζήτησε να μιλήσω για τους συναδέλφους. Αν πούμε μόνο δύο λεπτά θα σας δώσουμε τα αρνητικά στοιχεία, τα τέσσερα και τα θετικά. Λοιπόν, τέσσερα λεπτά θετικά. Γίνονται σαφέ αναφορέ στη βιώσιμη ανάπτυξη, του στόχου και τη Συμφωνία των Παρισίων. Ευπρόσδεκτα αυτά, θα επεκταθούμε από αυτόν. Δεύτερον, θετικό, διαγραφή τη ρήτρα να μεταφερθούν χρήματα από την πολιτική συνοχή σε αυτό το μέσο. Υποστηρίζουμε αυτή τη θέση, συνάδει με την οικονομική αντοχή. Δεν θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική η στόχη τεθέντε τρίτων, αλλαγή των ονομάτων, στον τη μεταρρύθμιση, το εργαλείο μεταρρύθμιση συγκλήσεω και το μέσο για τη διευκόλυνση τη ένταξη στην Ευρωζώνη είναι ενδιαφέρον συμβολικά, λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, συνέπειε των μεταρρυθμίσεων που έχει χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα. Κάποιε μεταρρυθμίσεις, αν χρηματοδοτηθούν σε ένα κάτω μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά σε άλλο κάτω και θα πρέπει να ενθαρρύνει το μέσο ε, κάποιες μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν προβλήματα γειτονική. Για τη σύγκληση πρέπει να αυξηθεί η ακρίβεια όσον αφορά τα κριτήρια σύγκληση και την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών που απαιτούνται για την συμμετοχή στην Ευρωζώνη. Όμω. Θα κάνουμε προτάσει για διεύρυνση των επιλεξίμων ρυθμίσεων, γιατί επιτυχή προσχώρηση στην Ευρωζώνη απαιτεί κάτι παραπάνω από ονομαστική προσαρμογή και νομική εφαρμογή, ε, ευθυγράμμιση. Μετά το θέμα τη διακυβέρνηση, ο συγγητή άλλαξε την αρχική εφαρμογή σε κατεξουδότηση πράξη, ώστε να υπάρχει σε εφαρμοστική μάλλον ε, ε, διάταξη. Πρόβλημα. Δεν αλλάγεται η κλίδα κατανομή. Υπάρχει έλλειψη αλλαγή και είναι προτεραιότητα για την ομάδα μας ούτε από σύνδεση μεταξύ RSP και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, άρθρο 8 παραμένει αμετάβλητο, ενώ είναι από τα πιο προβληματικά άρθρα, χωρί να τροποποιηθεί το σχέδιο εκθέσεως, έχασε την ευκαιρία να πετύχει του στόχου, του στόχου των Παρισίων και του κοινωνικού πυλώνα τη Ενώση στα πλαίσια των, ε, του προγράμματο υποστηρίξεων μεταρρυθμίσεων. Δεν αλλάζουν επίση τα στοιχεία. Ίσως λόγω του, της εκθέσεως ε, για, την, για το πολιτέ κοινωνικό πλαίσιο μετά το 2020 δεν υπάρχει σωστή ισορροπία για το μέσο αυτό. Μετά ο ρόλος του ανεξαρτήτου ε, δημοσιονομικού Ινστιτούτου. Ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς και θα πρέπει να δίνει δημοσιονομική ανάλυση και να δίνει αριθμούς χωρίς να αναφέρεται σε επιλογές πολιτικών. Και επιμένω ότι οι περισσότεροι ανεξάρτητοι οικονομικοί ε, φορείς Ινστιτούτο καθοδηγούνται από μόνο μία οικονομική θεωρία, την νεοκλασική οικονομική θεωρία, που είναι στα μοντέλα που τελικά δεν λειτουργούν και είναι εσφαλμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία λεπτά, είδατε. Ευχαριστώ που χρησιμοποίησατε μόνο τρία λεπτά. Γκουε, Econ Budget, υπάρχει κανείς. Κανείς. EFDD. Ο κ. Βάλλη, για δύο λεπτά. Γενικά, θα ήταν χρήσιμο να στηρίξουμε αυτέ τι διορθωτικέ αλλαγέ. Βιώσιμε μεταρρυθμίσει. οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, υπέρ τη ανάπτυξη. Τα κράτη-μέλη έτσι να μπορέσουν να πάνε σε αυτή την κατεύθυνση και να γίνουν αυτά προτεραιότητες για τα κρατημέλη. Και επίσης θα πρέπει να βρούμε ποια θα είναι τα κριτήρια του παραδεκτού, κάτι το οποίο να συμβαδίζει με τους στόχους της Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει το πρόγραμμα να στηρίζει τις ε, μεταρρυθμίσεις που θα έχουν σχέση με αυτά που είπαμε. Με εδαφική, βιώσιμη ανάπτυξη, ε, πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ε, νομιμότητα, κατά της απάτης, απασχόληση με επιτικές συνθήκες, ε, ισότητα κοινωνική κλπ. Σωστά το είπαν μέχρι τώρα οι που είναι εδώ, αλλά θα πρέπει να τα ξαναπούμε και να τα θωρακίσουμε περισσότερο στο μέλλον. Οπότε το πρόγραμμα αυτό θα, θα πρέπει να βοηθήσει εκεί που έχουν χτυπηθεί οι μισθοί και η απασχόληση. Γιατί αυτά είναι δυσκολίες που θα, θα τις βρούμε μπροστά μας όσον αφορά τη διαχείριση ε, της διαδρομής που οδηγεί σε σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε φυσικά θα ξεσηκωθεί ο κόσμος εάν έχουμε περικοπή των μισθών και Οπότε χρειάζεται κάποια αξιολόγηση εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Δεν συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δική αξιολόγηση όσον αφορά τη, τις εθνικές δημοσιονομικές αρχές. Και δεν θέλουμε επίσης να υπάρχει κάποια πειθαρχία κεντροκατευθυνόμενη γιατί αυτή οδηγεί σε ανισορροπίες. Ευχαριστούμε κύριε Βάλλη. Όμως από το ENF δεν παρισταται κανείς. Ούτε ζητεί κάποιος άλλος τον λόγο. Άρα να δώσουμε τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο λεπτά. Um, Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη όσων μας υπεστήριξαν για την πρότασή μας να σας πω δύο λόγια για αυτή την διευκόλυνση της σύγκλησης και το πεδίο εφαρμογή Όλα αυτά γίνονται για να βοηθήσουμε τα κρατημήλια τόσο ώστε να μην έχουμε μόνο τα κριτήρια της ονομαστικής σύγκλησης. Και έτσι να μπορέσουν να πληρώνουν τα κριτήρια και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Έχουμε και τις επιπλέον προτάσεις ζητούμε περισσότερα όσον αφορά τα μέτρα σύγκλησης κόστος, όφελος στη μελέτη αυτή. Ε, να το διευκολύνουν τα κρατημέλη, να μην είναι τόσο δύσκολη η υποβολή προγράμματος. Για την ε, απαλυσή της μεταφορά πόρων, ε, περίεργο αυτό, γιατί να έχουμε κάποιες χώρες που ε, έχουν χρησιμοποιήσει αυτήν την δυνατότητα της τεχνικής αρρωγής. Θα πρέπει όλα αυτά να είναι απλά και λειτουργικά. Αλλιώς δεν γίνεται να επιτευχθεί συμφωνία. Για την ιδιοποίηση τώρα της μεταρρύθμισης, ε βέβαια, αυτό θέλουμε να κάνουμε με την πρότασή μας. Μα μόνο αν θέλει το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει την πρότασή του. Οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις επίσης καλύπτονται σε αυτή τη μεταρρύθμιση θα είναι ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και επίσης, να δούμε πώς η πολιτική σύνοχη θα καλυφθεί από το κόστος των επενδύσεων για να προχωρήσουμε στην διαρθρωτική μεταρρύθμιση αυτά. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ε, έχουμε προχωρήσει παραπάνω γρήγορα από ό,τι προβλεπόταν. Επομένω, τώρα μπορούν οι συν να έχουν τρία λεπτά εκάστη. Well, thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα προσπαθήσω να προηγηθώ στα δύο λεπτά γιατί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε κάποια θέματα, να δώσω μία απάντηση προ το ΕΛΚ και ενδεχομένω και σε ό,τι αφορά του πράσινου. για τα ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθούν νέα όργανα, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε να εργαστούμε επί μια τέτοια βάσης σε ό,τι αφορά τα κρατή μέλη τη Ευρωζώνη και κάτι άλλο που ήθελα να σχολιάσω για το ECR και το σχόλιο του κυρίου Λούκα για τον ηθικό κίνδυνο. Σύμφωνο απόλυτα με τα σχόλιά του. Γι' αυτό και θα πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή και προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Προσβλέπω λοιπόν και στη μελλοντική συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καρτία Ζαβάλ. Για να προσθέσω γρήγορα να απαντήσω πρώτα πρώτα όσον αφορά το κριτήριο της ε, διανομής, κατανομής, γιατί αναφέρθηκε από πολλές πολιτικές ομάδες. Κάναμε μία απόπειρα με την ε, συμφωνία να αλλάξει το κριτήριο, αλλά δεν τα καταφέραμε να τα βρούμε. Δεν είναι είναι λογικό κριτήριο. Ο πληθυσμό δεν μπορεί να είναι το μόνο κριτήριο για την κατανομή των πόρων. Θα προσπαθήσουμε με νέε προτάσεις. Α, δούμε. Να πάμε στην κατανομή όπως στην πολιτική συνοχή ή σε κάτι άλλο. Λογικό. Όσον αφορά τώρα τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων, Όχι κύριε Λαμασούρ, δεν έχουμε μπει στην ουσία. Είπαμε να δώσουμε μια παράταση ενό έτου. Αυτό θα περιβάλλει με ασφάλεια τη μεταρρύθμιση και τη συνέχισή τους. Αλλά εντάξει, αυτό που λέτε κύριε Λαμασούρ, μπορούμε να το περιλάβουμε. Για την ρεσιμότητα και το κράτος δικαίου Είναι και άλλε επιτροπέ συναρμοδίε και ξαφνικά όλοι θέλουν να βάλουν ένα άρθρο για το κράτο δικαίου. Ε, δεν χρειάζεται. Α, συνεισηγητή μου για το κράτο δικαίου είναι και ο Σαραβαμά που μα προεδρεύει τώρα. Όλα τα προγράμματα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσουν από, από τη, την κρυσάρα του, του, αυτού του κανονισμού για το κράτος δικαίου. Όπω και όλα και όλα. Άρα Όλα τα προγράμματα πρέπει να συμβαδίζουν με αυτή την αρχή. Δύο σχόλια. Όσον αφορά τον ηθικό κίνδυνο, ότι πρέπει να συζητηθεί επί τη τραπέζη, να τεθεί. Ναι, ναι, ναι, σε κάποιε πολιτικέ ομάδε αρέσει πάρα πολύ, αλλά μιλάμε για τέτοια ποσά. Μιλάμε για τέτοια ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε χώρα με αυτό το πρόγραμμα. Και έτσι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο όσον αφορά την πάυση των μεταρρυθμίσεων όσο υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ. Ε, για οποιοδήποτε προπολισμό οποιασδήποτε χώρα είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κίνδυνος για το front load. Καμία πρόταση δεν υπάρχει, προκαταβολής. Η δε πολιτική μας ομάδα λέει ότι όταν αυτά τα χρήματα εκταμιευτούν όχι μόνο θα έχει τελειώσει η μεταρρύθμιση, θα έχει ξεχαστεί κιόλα. Άρα τι front loading. Πάνω αυτά. Και επίσης όσον αφορά τα όσα είπαν οι πράσινοι για το κοινωνικό πυλώνα, για το COP21, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ένα τελευταίο τώρα για το ΠΠ και τους πράσινους για, τους, ε, για τα κονδύλια αύξηση και να πάμε σε χώρες εκτός Ευρωζώνης. Μιλάμε για 22 δις. Πού να φτάσουν αυτά. Δεν το νομίζω. Υπερβάλλουν εδώ οι πράσινοι. Και όχι μόνο για το κριτήριο του πληθυσμού, με οποιοδήποτε κριτήριο. Καλύτερα να διπλασιαστεί η προοικοδότηση, αλλά δεν ισχύει αυτό τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Γκρατιασάλη για το κράτος δικαίου. Πράγματι σε αυτή την νομοθεσία όπως και σε άλλες. Είναι πολύ δημοφιλές θέμα το κράτος δικαίου. Πολλά έχουν υποθεί για την καλύτερη νομοθεσία. Ας δώσουμε το καλό παράδειγμα λοιπόν και μέρους των, της Επιτροπής Οικονομικών και Ζωνοπτικών Θεμάτων και Προϋπολογισμών και να αποφύγουμε κείμενα που δεν είναι απαραίτητα. Να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 3 ώρα το μεσημέρι, στις 15 Ιανουαρίου 2019, η ψηφοφορία στην Budget Kekon ή 20-21 Φεβρουαρίου του 2019. Για τα διάφορα δεν υπάρχουν διάφορα προς Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα όταν καθοριστεί. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα και εδώ ολοκληρώσαμε συνεδρίαση πέντε λεπτά νωρίτερα. Ευχαριστώ.